Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν οι άνθρωποι για κάτι το οποίο πριν ήταν δωρεάν. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρέντεργκαστ. Έκθεση Bradborn για το μέλλον των περιφερειακών αεροδρομίων. 94 του 2012. Τον λόγο έχει ο συγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που παρουσιάζω την έκθεση πρωτοβουλίας για τις περιφερειακές αερομεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση αυτή βασίζεται στην αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που οι περιφερειακές ε, συνδέσεις, αεροπορικές συνδέσεις παίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την οικονομική ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επιβίωση των περιφερειών. Οι εταιρείε αυτές συνδέουν 150, ε, μάλλον ε, υπάρχουν εκατοντάδες ε, τέτοιες χιλιάδες συνδέσεις ανάμεσα σε μικρότερες πόλεις και δεν απομονώνονται περιοχές των κρατών μελών, διευρύνονται οι εταιρικές σχέσεις το εμπόριο, προωθούνται οι οικονομικές δραστηριότητες και μερικές φορές συνδέουν πράγματι ακραία περιφερικές ζώνες με ε, την υπηρετική χώρα. Παρ' όλα αυτά οι αερομεταφορές αυτές ε, έχουν λίγα περιθώρια κέρδους για σωστή λειτουργία, αντιμετωπίζουν προβλήματα από τη μικρή κίνηση, μερικές φορές από τις ε, καιρικέ συνθήκες πρέπει να μην υπάρχουν εμπόδια και πρέπει τα αεροδρόμια τα περιφερικά να αντιμετωπιστούν σαν ολοκληρωμένο τμήμα των ευρύτερων δικτύων των ευρωπαϊκών και όχι σαν κάτι το εξωτικό. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στην βιομηχανία έτσι ώστε να προωθήσει συνδυασμένες μορφές μεταφορών όπως ακριβώς ε, η η δυνατότητα έκδεσης πολλαπλών εισιτηρίων κτλ. Λοιπόν, οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν με τα προγράμματα ΚΕΣΑΡ όπως επίσης και με το πρόγραμμα για τους ενιαίους ευρωπαϊκούς ουρανούς, είναι απαραίτητα. Υπάρχουν αεροδρόμια τα οποία δεν λειτουργούν όσο θα μπορούσαν μέχρι τώρα και θα μπορούσαν να ελαφρύνουν τον συνοστισμό σε κεντρικό αεροδρόμια. Η ενθάρρυνση συνδέσεων από περιφέρεια σε περιφέρεια θα ελαφρύνει επίσης ε, τον συνοστισμό στα κεντρικά αεροδρόμια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να, να προσέξει ε, τις περιφέρειες οι οποίες κινδυνεύουν να απομονωθούν λόγω της έλλειψης οικονομικών κινήτρων. Επίσης ε, τίθεται και το θέμα της διαφάνειας της τιμολόγησης των ε, υπηρεσιών των αερομεταφορέων. Ε, επιβαρύνουν την αρχική τιμή και μερικές φορές κάποιες εταιρείες προσφέρουν την δυνατότητα στους πολίτες να πληρώνουν μέσω πιστοτικών καρτών χωρίς έτσι να υφίστανται επανειλημμένες επιβαρύνσεις φορολογικές και χωρίς να αναγκάζονται να εκδίδουν πολλαπλά εισιτήρια. Σχετικά με τις αποσκευές πρέπει να τεθεί ενιαίο ανώτατο βάρος για μέγεθος και το βάρος φυσικά πρέπει να είναι καθορισμένο το ανώτατο. Θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν από τον κανόνα της μίας τσάντας για είσοδο στο αεροσκάφος τα προϊόντα τα οποία πολλούνται στα καταστήματα των αερολιμένων. Η πρακτική η οποία ισχύει σήμερα δημιουργεί προβλήματα στα αεροδρόμια αυτά και αναγκάζει στην αύξηση των εισιτηρίων. Εν πάση περιπτώσει, οι αερομεταφορέ, οι περιφερικέ και τα περιφερειακά αεροδρόμια παίζουν ρυθμιστικό ρόλο στην οικονομία και στο ευρύτερο ε, δίκτυο μετακινήσεων. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθήσει να πάρει μέτρα έτσι ώστε να διευκολύνει τους καταναλωτές, τους ταξιδιώτες και τις υπηρεσίες. ευχαριστώ κύριε Περνάμε στο και έτσι Τον λόγο έχει ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά τα οποία είπε ο εισηγητής και τον συγχαίρω για την πρωτοβουλία του. Οπωσδήποτε τα περιφερειακά αεροδρόμια έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν στις μεταφορές και οπωσδήποτε πρέπει να συμπεριληφθούν στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Πρέπει να δούμε και τον κανόνα της μίας χειραποσκευής που είναι προβληματικός για τα μικρά αεροδρόμια. Είναι σημαντικό να ε, αποδίδουν οικονομικά τα μικρά αεροδρόμια και βεβαίως ε, προϋπήρχαν ε, κάποια από δρομολόγια θαλάσσια ή από κάποια δρομολόγια τρένων. Οπότε πρέπει να δούμε μια γενικότερη άποψη αλλά εάν έχουν γίνει άχρηστα κατά κάποιον τρόπο, δεν έχει νόημα να σπαταλάμε χρήμα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. ευχαριστώ, η κυρία Τσικάου. Ευχαριστώ η περιφερειακή αεροπορία είναι πολύ σημαντικό παράγοντα για να μπορούν να μετακινούνται οι πολίτε. Τα περιφερειακά αεροδρόμια είναι πολύ σημαντικά και για την εδαφική συνοχή και για την ανάπτυξη την οικονομική και την κοινωνική πολλών περιφερειών, περιφέρειες που μερικέ φορέ δεν έχουν άλλα μέσα μεταφορά. Η πολυτροπικότητα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική γιατί μόνο έτσι θα βελτιώσει την πρόσβαση στις διάφορες περιφέρειες και την ανάπτυξη του τουρισμού εκεί. Δυστυχώς τα περιφερειακά αεροδρόμια όμως είναι μακριά από τα αστικά κέντρα και πολύ συχνά δεν συνδέονται καλά με τις επίγες μεταφορές, με τις οδικές, με τους αεροδρόμους. Πρέπει λοιπόν η Επιτροπή να παρουσιάσει σχέδια για την βιώσιμη κινητικότητα. Να προβλέπετε μια αποτελεσματική αλυσίδα διαχείριση. Και πρέπει να υπάρχει και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των περιφερειακών αεροδρομίων και των αστικών κέντρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει του καλύτερου προσανατολισμού προκειμένου να έχουμε την καλύτερη δυνατόν εξέλιξη των αεροπορικών υπηρεσιών και να έχουν και τις υποδομές που πρέπει για να σεβαστούμε την πολυτροπικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φερέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χρειάζονται ευρύτερε στρατηγικές και τα περιφερειακά αεροδρόμια πρέπει μέσα σε αυτέ να εντάσσονται για την, ε, το ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξη. Πρέπει να βοηθήσουμε την καταπολέμηση των συμμετριών στην περιφέρεια. Χρειάζεται επίσης καλή σύνδεση με άλλους τρόπους μεταφοράς, θαλάσσιους, οδικές μεταφορές και να βελτιωθεί έτσι η κινητικότητα των ατόμων αλλά και των εμπορευμάτων, λαμβάνοντα υπόψη όμως και το περιβάλλον. Πρέπει να προσέξουμε πού θα δώσουμε τι θα υπογραμμίσουμε. Το συμφέρον πρέπει του κόσμου να υπογραμμίσουμε πάνω απ' όλα και πρέπει ό,τι ρυθμίσεις αποφασίσουμε η παρέμβαση και η κρατική ρύθμιση να λαμβάνουν υπόψη τους στην αγορά. Δυστυχώς έχουμε προχωρήσει σε κοινωνικό dumping όμως αυτό το τομέα με ένα επίπεδο πολύ χαμηλό ηθικών εργασίας. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πάσκο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Λόγω του ότι η Ευρώπη είναι πύκνο κατοικημένη και λόγω της βιομηχανικής παραγωγής έχουμε πολλά αεροδρόμια που διαφέρουν ε, από πλευράς ε, μεγέθους και υπηρεσιών. Πέρα από τα μεγάλα διεθνή αεροδρόμια, οι μεταφορές ε, ανθρώπων και εμπορευμάτων καλύπτονται από σημαντικά περιφερειακά αεροδρόμια που στηρίζουν την ενδοχώρα τους, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου η κινητικότητα των πολιτών έχει νέες διαστάσεις ε, σωστή διαχείριση των αερομεταφορών είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό σωστό είναι να δούμε τις ιδιαιτερότητες των περιφερειακών αεροδρομίων που λειτουργούν διαφορετικά από τους μεγάλους κόμβους, τους οποίους κυρίως αφορά η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Οι ιδιαιτερότητες λοιπόν των περιφερειακών αυτών αεροδρομίων πρέπει να ληφθούν υπόψη όπως προτείνει ο κ. Μπράντμπορν για να εξασφαλιστεί η σωστή τους λειτουργία στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Πέρκερ. Ευχαριστώ. Με την έκθεση αυτή τονίζουμε την ιδιαίτερη σημασία των περιφερειακών αεροδρομίων αφενός ως ε, συγκοινωνιακών κόμβων και αφετέρου ως ε, σημαντικής οικονομικής δραστηριότητας της περιφερειάς και για την Ένωση γενικά. Για να ενισχύσουμε αυτά τα αεροδρόμια θα ήθελα να αναφέρω τρία σημεία. Πρώτον, η σύνδεση με άλλα μεταφορικά μέσα. Δεύτερον, τα περιφερειακά αεροδρόμια πρέπει να συνδεθούν πιο πολύ μεταξύ τους και τρίτον, αν υπάρχουν στενοποί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικά αεροδρόμια. Επίσης, πρέπει να είναι ξεκάθαρο πως τα περιφερειακά αεροδρόμια δεν πρέπει να γίνουν μνημεία ε, τοπικών πολιτικών ε, αλλά πρέπει να μπορούν να αποδίδουν οικονομικά, να μην είναι ε, ελληματικά. Τέλος, να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Μπράντον, για την συνεργασία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Πίρκερ. Η κυρία Πρέντεργκαστ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε τα τέσσερα περιφερειακά αεροδρόμια στην δική μου εκλογική περιφέρεια στην Ιρλανδία θα επωφεληθούν νομίζω από την έκθεση αυτή. Καλωσορίζω ε, την παρατήρηση για, την, ε, για τον κανόνα της μίας χειραποσκευής η οποία ωφελεί τις αεροπορικές εταιρείε, αλλά βλάπτει τα αεροδρόμια γιατί βασίζονται σε λιανικές πωλήσει και πωλήσει τροφίμων πολλά από αυτά. Οπότε αν έχουν μόνο μία αποσκευή επιβάτες δεν μπορούν να ε, αγοράσουν πράγματα επιβάτες. Θα ήθελα επίσης ε, επί τη ευκαιρία να τονίσω τη σημερινή απόφαση της ε, Ιρλανδικής κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει το αεροδρόμιο Σάνων. Ελπίζω με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τέλος, ε, ο κύριος Νικολέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση Bradborn είναι ε, πολύ καλή για διάφορους λόγους. Πρώτον ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεώρησει την οδηγία η οποία καθορίζει ε, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να λάβει επιδοτήσεις ένας αερολιμένας, ο οποίος μπορεί να ε, χρηματοδοτηθεί εφόσον εξυπηρετεί άνω των 500.000 επιβατών κατέτος. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Η πολιτική η οποία ακολουθείται επίσης σε σχέση με τις χειραποσκευές είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει επίσης στα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών να ενταχθούν πάρα πολύ περιφερειακοί αερολιμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα οδηγήσει στην περαιτέρω οικονομική ανάκαμψη σχετικά με την με την αιτιολογική σκέψη 1 σχετικά με την εγκύτητα ενός αερολιμένος με την πρωτεύουσα ε, θα πρέπει οι κανόνες που καθορίζουν ε, το επίπεδο των αεροδρομίων να αναθεωρηθούν. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία και της ΔΙΑΗ. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Τουκιούχτη για να κλείσει η συζήτηση. Thank uh, uh, Ευχαριστώ. Πρόεδρε, εξότιμοι ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ για την έκθεση του κυρίου Μπράντμπορν για το μέλος των περιφερειακών αεροδρομίων και της αεροπορικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πακέτο πρωτοβουλίας υποβλήθηκε το Δεκέμβριο που μας πέρασε προκειμένου τα αεροδρόμια να είναι μια ιστορία επιτυχής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ουρανού. Χάρη σε αυτό, πολλοί νέοι δρόμοι έχουν φτιαχτεί, έχουν διπλασιαστεί βασικά τα τελευταία χρόνια. Τα περιφερικά αεροδρόμια συνδέουν τους πολίτες μεταξύ τους και έχει αλλάξει το τοπίο των περιφερειακών αεροδρομίων. Υπάρχουν τα τσάρτες πρώτα απ' όλα, τα οποία ε, πηγαίνουν τους τουρίστες σε νέους προορισμούς. Υπάρχει ένας ε, τομέας επίσης που προσφέρει έτσι ανάπτυξη και στις περιφέρειες. Τώρα για τα κύρια στοιχεία πολιτικής που αναφέρονται στην έκθεση του εισηγητή. Οι Γενικέ Διευθύνσει της Επιτροπής μελετούν την ε, μεταρρύθμιση όσον αφορά τι κατευθυντήριε γραμμέ για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Ο ρόλος των περιφερειακών αεροδρομίων είναι η εδαφική συνοχή και η διασύνδεση των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αποτελεί μια προτεραιότητα. Δεν μπορούμε όμως να γνωρίσουμε συγχρόνως το ότι ο αθέμητος ε, ανταγωνισμός μέσω κρατικών ε, επιχορηγήσεων στρεβλώνει πράγματι κάθε επιχορήγηση κρατική των ανταγωνισμό. Η έκθεσή σας σίγουρα θα ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη στα πλαίσια της αναθεώρησης που κάνουμε. Το θέμα του περιορισμού των χειραποσκευών με την μία επιτρεπόμενη χειραποσκευή. Οι επιβάτες είναι αλήθεια ότι κάθε φορά που αντιμετωπίζουν τέτοιους περιορισμούς όταν φτάνουν στο αεροδρόμιο μπερδεύονται. Η Επιτροπή μελετάει το θέμα στα πλαίσια της έκθεσης αντικτύπου που κάνει για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών ε, ε, εταιριών 261-2004. Όσον αφορά τώρα το λιανικό σκέλος, έχει να κάνει με τις σχέσεις των επιχειρήσεων μεταξύ τους, με τον ανταγωνισμό. Αν υπάρχουν θέματα ανταγωνισμού, αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά όχι να αλλάξουμε την νομοθεσία που προστατεύει τους επιβάτες. Υπάρχει και η προτινόμενη αλλαγή στο, στη ρύθμιση για τα σλότς. Ο Επίτροπος Κάλλας λέει ότι ο στόχος δεν είναι βέβαια να αποκλείσουμε από την αγορά τα περιφερειακά αεροδρόμια, αντίθετα να αυξήσουμε την ε, δυνατότητα υποδοχής κοινού. Το θέμα του πληστηριασμού των σλότς έχει αποκλειστεί πάντως, γιατί πιστεύουμε ότι δεν είναι ότι καλύτερο. Συνεχίζονται πάντως συζητήσεις και στο Συμβούλιο και εδώ στο Κοινοβούλιο. Το θέμα της πολυτροπικότητας τώρα επίσης είναι στην καρδιά της πολιτικής μας μεταφορών. Τα περιφερειακά αεροδρόμια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο μέλλον μέσα στα πλαίσια της πολιτικής μας μεταφορών. Είναι όντως καθήκον των διευρωπαϊκών δικτύων να λάβουν υπόψη τους και τα περιφερειακά αεροδρόμια. Χρειάζεται όμως να λάβουμε υπόψη μας τις νέες τεχνολογίες. Η ιδέα ενός πανευρωπαϊκού συστήματος εισιτηρίων λοιπά είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου. Η Επιτροπή επίσης εξετάζει την πρακτική ορισμένων αεροπορικών εταιριών να επιβάλλουν τέλη ή επιπλέον κόστος στην περίπτωση που πληρώνουν τα εισιτηριά τους, για παράδειγμα, επιβάτες με επιστοτική κάρτα. Κάνουμε μία μελέτη για να δούμε κατά πόσο όλα αυτά είναι συμβατά με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. πρέπει να μπορεί κανείς να πληρώνει με τον τρόπο που θέλει. Πρέπει να συζητήσουμε και με τις αρχές των κρατών μελών για να δούμε τι τελικά μπορεί να επιτρέπεται και τι όχι. Τα αεροδρόμια πάντως είναι πολύ σημαντικά για την Ευρώπη και αποτελούν και ε, μηχανισμούς ανάπτυξης. Συνδέουν επίσης τις άκρος περιφερειακές περιοχές της Ευρώπης με το κέντρο. Θα ολοκληρώσω ευχαριστώντας σας για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση που άκουσα για αυτό το σημαντικό θέμα. Η Επιτροπή περιμένει τη συνέχεια. Έχουν οι συζητήσεις για ολόκληρο το πακέτο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ κύριε Ντεγκύχ. Τελείωσε η συζήτηση. Να σας υπενθυμίσω πως η έκθεση του κυρίου Μπράντμπορν έχει γίνει στην έκθεση έχει γίνει ένα λάθος. Υπάρχει διόρθωση σε όλες τις γλώσσες. Η ψηφοφορία αύριο στις 11.30. Η, η συνεδρία θα επαναληφθεί αύριο το πρωί. Η διάταξη έχει δημοσιευτεί, είναι στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλό σας βράδυ.